Panie Przewodniczący! Witam Państwa bardzo serdecznie. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με τις εργασίες μας. Τα χθεσινά πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα είναι ήδη διαθέσιμα. Τώρα. Έχω δήλωση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που υποβλήθηκε όσον αφορά τις οικονομικές γραμμές. Πρόκειται για το άνοιγμα της